ξεκάθαρα και απερίφραστα να ε, επιβεβαιώσουμε τις προτεραιότητες μας για μια εναρμονισμένη διαδικασία στον τομέα αυτών. Η συζήτηση έληξε, η ψηφοφορία θα διεξαθεί την Τετάρτη στις 12. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Lightfried, έλεγχος των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης. Το λόγο έχει ο εισηγητής μας, ο κύριος Lightfried, για τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως και σε σχέση με την έκθεση για τις ε, άδειες ε, εξαγωγής ε, ειδών διπλής χρήσης και σε σχέση με το τις συνολικές πτυχές όλων που θα έπρεπε συνολικά να καλυφθούν και για την οικονομική πρακτική που ακολουθείτε, που πολλές φορές ε, βρίσκεται, ας το πω έτσι, ε, υπό ένα καθεστώς ε, υποψίας που επισκιάζει αυτές τις διαδικασίες θα πρέπει πανευρωπαϊκά να μπορέσουν να ρυθμιστούν αυτά τα θέματα. Πρόκειται για διευκόλυνση αδειών εξαγωγής για προϊόντα που και σε πολιτικό επίπεδο αλλά αστικό επίπεδο και σε στρατιωτικό επίπεδο μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πρόκειται για χημικές ουσίες, πρόκειται για εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και πρόκειται και έχουμε συζητήσει και για λογισμικό και για μέρη και τμήματα λογισμικού. Εδώ είναι σημαντικό πιστεύω να διαφοροποιήσουμε και να πούμε ότι οι διαφορετικοί κανόνες και κανονισμοί που υπάρχουν στα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταλήξουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Να μπορέσουμε να καθορίσουμε αυτές τις ενιαίες διαδικασίες και να είναι πιο διαφανείς αυτές οι διαδικασίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαφανείας. Και σε αυτή την έκθεση ίσως από τις πρώτες φορές έχουμε και την εφαρμογή των επιπτώσεων της συνθήκης της Λισαβόνας που μπορούμε να δούμε τις επιπτώσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά είχε υποβάλει αυτή την πρόταση στο Συμβούλιο θεωρώντας ότι μέχρι την ολοκλήρωση της ε, συνθήκης ε, της Λισαβόνας θα μπορούσε να ε, ευδοκιμήσει. Δεν συνέβη αυτό. Κατέληξε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι καλό το ότι κατέληξε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι βλέπουμε κάποια πράγματα διαφορετικά από το Συμβούλιο και θέλουμε να παρέμβουμε καταφέραμε σε σχέση με τις νομικές επιπλοκές ε, που ε, πέρευσαν από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα και κινηθήκαμε σε ένα πλαίσιο νομικής ε, βεβαιότητας και ασφάλειας. Και εμείς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο ουσιαστικά στα περισσότερα πράγματα συμφωνούμε μέχρι κάποιες λεπτομέρειες και σε σχέση και με το Συμβούλιο επίσης. Πρόκειται για το ζήτημα ε, θα πρέπει να εγκρίνονται οι εξαγωγές ε, όταν θα έχουν γίνει ή πριν ε, συμβούν, πριν γίνουν. Και είναι λογικό πιστεύω για λόγους ασφάλειας, για λόγους σωστής εποπτείας και διαφάνειας να πούμε ότι πρώτα πρέπει να υπάρχει η άδεια προτού εξαχθεί κάτι το οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο και όχι στη συνέχεια εκ των υστέρων και γι' αυτό θα πρέπει να ε, καταφέρουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο να δράσουμε, γιατί διαφορετικά δεν θα είμαστε αποτελεσματικοί. Είναι η περίφημη περιβόητη συζήτηση εξ post ή εξ ante, εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων, σε σχέση με την αδειοδότηση για τέτοιου είδους εξαγωγές. Εκεί όπου συμφωνούμε όλοι μας, αλλά δεν συμφωνούμε με το Συμβούλιο, είναι το θέμα της διαφάνειας. Εγώ πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε όπως και αν επιληθεί το πρόβλημα, είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε, να γνωρίζουμε τι εγκρίθηκε, προς ε, ποια χώρα και με ποιον αποδέκτη, γιατί πρέπει να μεριμνήσουμε τα πράγματα να λειτουργούν σωστά μέσα σε ένα σωστό πλαίσιο. Και γνωρίζουμε ότι σε σχέση με τις ε, συζητήσεις που διεξάγονται για τις εξαγωγές, ε, πρέπει να, να έχουμε υπόψη ποιοι είναι οι τελικοί αποδέκτες και να αποφύγουμε καταχρήσεις και θα πρέπει να μεριμνήσουμε για την τελική χρήση να είναι η σωστή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Χαίρομαι ήδη για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Επιτροπής, η Επίτροπος κυρία Μάλστρομ έχει το λόγο. Yes, thank you, Mr. President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Σιγητά. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κάθε μέρα βρισκόνται σε μια σχέση ανταγωνισμού, σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό και προκλητικό παγκόσμιο περιβάλλον. Άρα λοιπόν πρέπει και ο χρόνος αλλά και οι τιμές, η ποιότητα, όπως και η ποιότητα να ε, υπολογίζονται. Χρειάζεται ειδική διαδικασία για χορήγηση άδεια για τα προϊόντα διπλή χρήση. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία θεμητά χρησιμοποιούνται σε μεγάλη γκάμα τομέων, είτε πρόκειται για την αεροβιομηχανία, είτε πρόκειται για τη χημική βιομηχανία ή την κατασκευαστική. Ελέγχονται όμω διότι μπορεί να έχουν χρήση και σε στρατιωτικου σκοπους σκοπούς. Ορισμένα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν ειδικέ διευκολύνσεις για του εξαγωγείς του με γενικέ άδειες που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις των κρατών μελών αυτών να εξάγουν αυτά τα προϊόντα διπλής χρήσης με ως το δυνατόν περιορισμένο γραφειοκρατικό ε, κόστος. Έτσι λοιπόν το 2009 θεσπίστηκε η πρόταση για την επέκταση αυτών των διευκολύνσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γενική άδεια εξαγωγή έχει σαν στόχο να επιτρέψει εξαγωγή όλων των κρατών μελών να δρέψουν τους καρπούς ε, αυτής της ε, άδεια για τα προϊόντα διπλής χρήσης και πάνω απ' όλα τη δυνατότητα να τα παρουσιάζουν και σε ε, εκθέσεις Πλουστεύεται λοιπόν ε, η εξαγωγή τους ε, και για τα προϊόντα των τηλεπικοινωνιών για ορισμένα χημικά στατικά. Ορισμένα τα κράτη-μέλη επίση θα μπορούν ε, του περιορισμένου του πόρου να του επικεντρώσουν από την άλλη πλευρά σε συναλλαγέ όπου πράγματι εντοπίζονται κάποιοι κίνδυνοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση πολλέ φορέ ακούει διαμαρτυρίε από τον κλάδο για κάποιε συναλλαγέ οι οποίε ελέγχονται σε ορισμένα κράτη-μέλη ενώ από άλλα κράτη-μέλη έχουν λάβει το πράσινο φω. Και έτσι προσπαθούμε να εκμηδενήσουμε αυτές τις ανισότητες σε μια εσωτερική αγορά. Μην ξεχνάμε επίση ότι και οι μεγάλοι ανταγωνιστέ μα έχουν μια ενιαία στάση στην, στον έλεγχο αυτών των εξαγωγών και θα πρέπει να μείνουμε πίσω. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Λάικτφριντ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση. Σα ακολουθεί τον ορθό δρόμο και ε, συνάδει νομίζω με την πρόταση Επιτροπή εκ μέρους Επιτροπής των Εξωτερικών αλλά και με, την, ε, με το χρόνο που έχει ως ομιλητής των Πρασίνων ο κ. Πιτσικόφερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα θέμα που σχετίζεται και με το εμπόριο αλλά και με την ασφάλεια. Έχουμε να κάνουμε τα προϊόντα διπλή χρήση που μπορούν δηλαδή και να εξυπηρετήσουν μια χρήση μη στρατιωτική αλλά και ταυτόχρονα να αξιοποιηθούν σε μια μάλλον ευαίσθητη, για να μην πω επικίνδυνη χρήση που έχει να κάνει με την ασφάλεια, στρατιωτική χρήση δηλαδή. Υπάρχουν ε, ορισμένε περιπτώσει όπω παραδείγμα το Υπουργείο Οικονομικών τη Γερμανία όπου δηλώνεται και παραθέτω ότι, μη, ότι πρόκειται για μη κρίσιμα αγαθά. Αυτό είναι σφαλμένο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις ε, κοινοβουλευτικές του επιτροπές έχει τοποθετηθεί αντίθετα μέχρι τώρα σε αυτή την δήλωση. Ως εκπρόσωπος λοιπόν της Επιτροπής των Εξωτερικών και της Επιτροπής για την ε, Άμυνα και την Ασφάλεια, που Επιτροπή για την Άμυνα και την Ασφάλεια, ήθελα να πω ότι έχουμε λάβει μια σαφέστατη θέση και έχουμε ε, διεκδικήσει σαφείς μηχανισμούς έλεγχου. Απευθύνω λοιπόν έκκληση προς τους συναδέλφους να ακολουθήσουν τις προτάσεις των δύο επιτροπών, της Επιτροπής των Εξωτερικών και της Επιτροπής ε, ε, για την Άμυνα και την Ασφάλεια και κυρίως να ακολουθήσουν την πρόταση του εισηγητή για τους ελέγχους. Εδώ έχουμε το κύριο ζήτημα αντιπαράθεσης που παραμένει ακόμη εκρεμές οι εκ των υστέρων δηλαδή έλεγχοι, που ενδεχομένως να εισάγουν λιγότερη ασφάλεια. Όμως εμείς θέλουμε περισσότερη ασφάλεια και για τον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και για τον εταίρο μας ε, τρίτο κράτος μέλος ή για, το, τρίτο κράτος ή για τον εμπορικό μας εταίρο. Δεν θέλουμε δηλαδή η αρχή που έχουν ακολουθήσει η Επιτροπή ΑΦΕΤ αλλά και η Επιτροπή του Εθνούς Εμπορίου του προηγούμενου ελέγχου, του προκαταρκτικού ελέγχου, να αντικατασταθεί από έναν εκ έλεγχο. Υπάρχουν κράτη όπως ε, οι κάτω και τελειώνω πρόεδρε, τα οποία δηλώνουν ρητά ότι δεν θα πρέπει να ακολουθείται αυτή η λύση. Και πιστεύω ότι προς το συμφέρον των πολιτών μας θα ήταν να ακολουθήσει η Ολομέλεια της προτάσεις των Επιτροπών. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, πρώτα και το Λαϊκό Κόμμα, η κυρία Κιώστιγκερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, ο κανονισμός για τη διτή χρήση προβλέπει γενικές άδειες για την εξαγωγή τέτοιων αγαθών και ειδών που εξάγονται σε τρίτες ε, χώρες ε, και υλοποιούν ανταποκρίνονται στους στόχους εξαγωγής. Αυτές οι γενικές άδειες θα πρέπει για τους εξαγωγείς ε, και μικρομεσαίους επιχειρηματίες να διασφαλίζουν ένα πλαίσιο ασφάλειας σχεδιασμού θα πρέπει να διευκολύνονται οι εξαγωγεί ε, από πλευρά τη Ευρώπη ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά του. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η καταλεπτόσα ε, αναφορά και οι ε, διαδικασίες που θα ισχύουν για αυτές τις εξαγωγές δεν είναι διευκόλυνση αλλά επιβάρυνση. Χωρίς αμφιβολία πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εξαγωγές που υφίστανται αυτή τη διτή χρήση θα είναι ασφαλείς και δεν θα αποτελούν κίνδυνο. Και τώρα, σε σχέση με το, την, την υπερβολική δαπάνη που δημιουργείται, η υπερβολική ε, γραφειοκρατική επιβάρυνση. Μπορούμε να αναφέρουμε για παράδειγμα μια ε, υπηρεσία ε, που παράγει τέτοιου είδους μηχανικά αγαθά για που θα πρέπει με τις επιβαρημένες αυτές προδιαγραφές για την εξαγωγή να μπορεί να λειτουργεί και να εξάγει. Αυτό ισχύει επίσης και για τον κώδικα εξαγωγής. Όταν έχουμε τέτοιου είδους διαδικασίες και έχουμε ασάφειες όσον αφορά τις διατυπώσεις, τίθεται το ερώτημα της υπερβολικής γραφειοκρατικής επιβάρησης και δαπάνης. Είναι σημαντικό οι εμπλεκόμενοι να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης απόφασης. Όμως θα πρέπει να ακολουθείτε μια ρεαλιστική πρακτική όσον αφορά την λειτουργικότητα όλων αυτών. Η ασφάλεια χωρίς καμιά αμφιβολία πρέπει να πριτανεύει. Στο τέλος θέλω να αναφέρω ότι αυτός ο κανονισμός θα πρέπει να οδηγήσει στην μείωση της γραφειοκρατικής επιβάρησης. Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να διασφαλίσουμε την οικονομία μας που θα μπορέσει μέσα σε ένα πλαίσιο διευκολύνσεων να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος ε, Σούστας για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφό μας Λάιχφριντ για αυτή την τόσο τεχνική έκθεση με επιπτώσεις για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει μέτρα ελέγχου για τα προϊόντα διπλής χρήσης ε, μέσω προληπτικών μέτρων, μέτρων πρόληψης, καθώς επίσης και με τις, ε, την έκδοση αδειών και τα τε, ε, τελωνιακά μητρώα προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφύγει και να προλάβει την διάδοση όπλων και μάλιστα όπλων μαζικής καταστροφής. Όμως το καθεστώς από πλευρά της Ευρώπης πρέπει να είναι πιο διαφανές και πιο ε, δημοκρατικό. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα ασφαλές και αποτελεσματικό όσον αφορά τις ειδοποιήσεις ε, και καταχωρήσεις αυτών των εξαγωγών που θα πρέπει οι αναφορές να συλλέγονται, να καταχωρούνται σε μητρώα ώστε να αποφεύγουμε την διάδοση ε, ειδών και όπλων μαζικής καταστροφής. Για την ομάδα συντονισμού για τα προϊόντα διτής χρήσης πρέπει να υποβάλει μια ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διευκολύνεται η διαδικασία ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με την εφαρμογή την εφαρμογή του κανονισμού ελέγχου για τέτοιου είδους ε, προϊόντα διπλής χρήσης. Και επίσης πρέπει να υποβληθεί μια μελέτη ε, εκτιμήσεων και επιπτώσεων σε σχέση με τα μέτρα αυτά. Όσον αφορά τα, τις διεθνείς προδιαγραφές ελέγχου πρέπει να βελτιωθούν. Έτσι, οι κατάλογοι για τα προϊόντα αυτά πρέπει να επικαιροποιούνται διεθνώς, σε διεθνές επίπεδο και μετά για τη χρήση στο κοινοτικό επίπεδο να μπορούν να λειτουργήσουν και αυτό ε, επιθυμούμε να γίνεται με την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι χωρίς αυτή τη συμμετοχή, όπως προβλέπει η συνθήκη της Σαβώνας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρινάλντι για λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφοι κύριε Επίτροπε, ακόμα και σήμερα το πιο δύσκολο για τον έλεγχο του εμπόριου είναι το εμπόριο όπλων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που καθιστούν δύσκολο τον έλεγχο αυτό, μεταξύ των οποίων το να μπαίνουν στο εμπόριο όπλα εξαιρετικά επικίνδυνα, μάλλον εργαλεία εξαιρετικά επικίνδυνα που μπορούν εύκολα να γίνουν όπλα. Αυτά είναι τα εργαλεία διπλής χρήσης. Άλλο πρόβλημα είναι η κακοφωνία των ελέγχων που καθιστά δυσχερή τον έλεγχο. Όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε για το θέμα αυτό, η Επιτροπή μας ζητούσε να αλλάξουμε έναν κανονισμό του 2000. Εν τω μεταξύ, ανακλήθηκε ο κανονισμός αυτός και με την ίδια αναχρονιστική πρόταση έπρεπε να προχωρήσουμε στην ενθορήση της πιο πρόσφατης πρότασης του 9. Όταν μπήκαμε στον τριμερή διάλογο είχε έρθει μια νέα νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση εκ νέου του ίδιου κανονισμού. Άρα το, το πρώτο αίτημα, ε, σαφείς κανόνες χωρί, με διαφάνεια και απλή κανόνες για τους ε, εξαγωγείς είναι το βασικό μας αίτημα. Τέσσερις θέσεις για τις θέσεις των φιλελευθέρων. Πρώτον, εξαγωγές μικρής αξίας ζητούμε και εμείς θεωρούμε είμαστε πολύ επιφυλακτικοί μάλλον για το σύστημα αυτό. Το Κοινοβούλιο ήδη περιόρισε τη μέγιστη αξία από τις 5.000 στις 3.000 ευρώ και βέβαια άλλα, και άλλα κριτήρια. Ο κατάλογος των χωρών προορισμού είναι περιορισμένος. Κάτι το θέλουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το μήνυμα ωστόσο είναι ασφάλεια, όχι μόνο εμπόριο. Και στο θέμα αυτό θα εξεταστεί στον τρίλογο. Είμαστε υπέρ των, της πολιτικής των εκ των προτέρων κοινοποίησης με υποχρέωση καταχώρησης. Τρίτον, διαφάνεια σε μέγιστο βαθμό. το, το κείμενο προτείνει ε, σε ενδιαφερόμενες πλευρές όπως τα οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δυνατότητα παρέμβασης στις διάφορες, ενημέρωση για τις διάφορες φάσεις της απόφασης και μέσω ή έκθεση σχετικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριος Σόλτς για ένα λεπτό. ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, Ευχαριστώ ρητά τον εισηγητή Γιώργ Λάιχφριντ για τη δουλειά που έκανε η σύνταξη αυτή τη έκθεση και το εύχομαι εξ ονόματο τη ε, ε, ομάδα μου κάθε επιτυχία στι δυσχερεί ε, αυτέ τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο που δεν παρίσταται το Συμβούλιο. Θα ήθελα να αναφερθώ στι τροπολογίε τροπολογίες του ΕΛΚΑ που δεν βοηθούν τον εισηγητή αλλά σε σχέση με την ε, θέση του Κοινοβουλίου την αποδυναμώνουν. Οι τροπολογίες ε, στοχεύουν να διευκολύνουν τέτοιου είδους ε, εξαγωγές οπλικών αγαθών. Δεν υποστηρίζει αυτήν την τροπολογία η ομάδα μου. Δεύτερον, η ομάδα μου έχει σημαντικά προβλήματα, θέλω να πω, όταν πρόκειται για διτής χρήσεως ε, αγαθά και υπάρχει ο στόχος να αποκλείονται ε, τρίτες χώρες ε, για παράδειγμα σε σχέση με περιορισμούς για εξαρτήματα υπολογιστών έχουμε, γνωρίζουμε το τι μπορεί να γίνει σε σχέση με καταχρήσεις τέτοιων αγαθών dual use. Έχουμε διατυπώσει μια τροπολογία από πλευρά μα και προς το συμφέρον των αναπτυσσόμενων χωρών ζητώ να υποστηριχθεί αυτή η τροπολογία μας. Ευχαριστώ ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πυρηνικό υλικό, ε, χημικές ουσίες ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ειρηνικούς σκοπούς. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν εξοπλίσει χώρες όπως η Λιβύη, η Φερρυπίν, με υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, ασφαλώς για όπλα. Η Ιταλία, η Μάλτα και πολλές άλλες χώρες καταγράφονται ως οι ε, προμηθευτές του καθόλου του Καντάφη. Πρέπει λοιπόν να καταπολεμηθεί αυτό το εμπόριο και ολόκληρο ολόκληρη βιομηχανία όπλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τεθούν υπό πολύ αυστηρούς ελέγχους και όρους διαφάνειας. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ε, αμφιβάλλουμε και για το πόση χρησιμότητα μπορεί να έχει αυτή η νέα επανάσταση των smartphones στην Βόρεια Αφρική και για το πόσο χρήσιμη μπορεί να αποβεί τελικά. Για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε αυτή η νομοθεσία ως νομοθετική πράξη στοχεύει στη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αγαθά αστικής και στρατιωτικής χρήσης ε, για αεροπλάνα, για παράδειγμα φορτηγά και τα λοιπά. Και δεν πρόκειται άμεσα για αναφορά των όπλων και προϊόντων της οπλικής βιομηχανίας και αυτό είναι ίσως παραπλανητικό. Θα πρέπει άμεσα να αναφερόμαστε και να ε, ρυθμίσουμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είναι αυστηρές οι προδιαγραφές και να εναρμονίζονται. Και με Σουηδούς επιχειρηματίες έχω συζητήσει οι οποίοι σε σχέση με τέτοιου είδους εξαγωγές θα ε, πρέπει να πούμε ότι αντιμετωπίζουν ένα διαφορετικό πλαίσιο από ότι οι Γάλλοι για παράδειγμα. Για παράδειγμα σε σχέση με τις τηλεπικοινωνίες ε, και τον εξοπλισμό για τηλεπικοινωνίες ε, πρέπει εδώ να μην υπάρξει δυσλειτουργία λόγω γραφειοκρατικής επιβάρυνσης και πρόκειται για μια σωστή αναφορά και καταχώρηση τέτοιου είδους ε, περιπτώσεων και υπάρχει νόμιμο αίτημα και συμφέρον για να διεξάγονται τέτοιου είδους, ε, να εξάγονται τέτοιου είδους αγαθά. Θα πρέπει να γίνεται αυτή, να ακολουθείται αυτή η διαδικασία ε, εκ προημίου και να μπορεί να καλύπτεται και η διαδικασία ex post. Πρέπει πιο αυστηρά, με αυστηρότερα πλαίσια να είμαστε αποτελεσματικοί και να ρυθμίζουμε αυτά τα πράγματα, αλλά να διευκολύνουμε αντί να επιβαρύνουμε με γραφειοκρατική επιβάρυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Ζέμκε για ένα λεπτό. Ε, Jeśli można, chciałem bardzo, panie przewodniczący, podziękować za zabranie. Ευχαριστώ. Θα σε ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Ποιο είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς δεν έχουν τα ίδια κριτήρια όλες οι χώρες της Ένωσης για την εξαγωγή προϊόντων διπλής χρήσης. Πιστεύω ότι ο στόχος μας θα πρέπει να είναι αυτός. Οι χώρες της Ένωσης να ακολουθούν παρόμοια στάνταρτ σε ό,τι αφορά την παραγωγή προϊόντων διπλής χρήσης. Ο κανονισμός αυτός θα έπρεπε να επικεντρωθεί ιδίως σε ένα θέμα. Την ανάγκη περιορισμού της ανέλεγκτης και ανεξέλεγκτης διάδοσης του λογισμικού, ιδίως για νέες τεχνολογίες για νέα προγράμματα. Είναι σημαντικό να παρεμβαίνουμε μέσω του κανονισμού για να ε, καταπολεμήσουμε την κυβερνοπειρατεία. Ο κύριος Πάσκου. Το θέμα της έκθεσης έχει ε, διπλά ευαίσθητο χαρακτήρα και πολιτικό δηλαδή και οικονομικό και έχει να κάνει με την απαγόρευση της χρήσεως αυτών των, ε, μάλλον των εξαγωγών αυτών των προϊόντων διπλής χρήσεως ε, είναι πολύ ασαφές το πεδίο και υπάρχει η προσπάθεια να ε, κλείσουν κάποια παραθυράκια και να αποτραπεί το άνοιγμα κάποιων άλλων στο μέλλον. Για κάποιους είναι πολύ αυστηρό το καθεστώς, για κάποιους είναι πολύ αποδυναμωμένο και χρειάζεται περισσότερη και διαρκή αναθεώρηση. Εγώ ως μέλος σαφέτη υπέρ μιας διαρκούς και πολύ σοβαρής ενίσχυσης αυτού του συστήματος ε, και προκαταβολικού ελέγχου χάρη στη Λισαβόνα μπορούμε να βοηθήσουμε ως κοινοβούλιο και ο ρόλος μας θα πρέπει να ενισχυθεί, όχι να παραγνωριστεί. Ε, του Πρώτα ο κύριος Γιάρ για ένα λεπτό. Ε, um Ευχαριστώ. Όταν πρόκειται για την χορήγηση αδειών εξαγωγή ειδών διτή χρήση, όλοι συμφωνούμε, πιστεύω, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαίοι κανόνε πρέπει να εξευρεθούν να μην ακολουθούν διαφορετικέ διαδικασίε στα κράτη-μέλη και να μην οδηγούμαστε σε στρεβλώσει του ανταγωνισμού. Διότι τότε θα έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα από το ευκταίο. Και φυσικά ακούγονται όλα λογικά όταν λέμε ότι θέλουμε οι εξαγωγέ πριν από την εξαγωγή να εγκρίνονται και να διοδοτούνται. Θέλουμε να είναι υπό πλαίσιο διαφάνειας και μέσα σε ένα πλαίσιο ε, αποτελεσματικών ελέγχων Θέλω να υποστηρίξω τον συνάδελφο που είπε ότι χρειαζόμαστε φυσικά επίση ένα σύστημα που για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει θα είναι λειτουργικό και θα είναι εφικτό και θα μπορούν να το υπομισθούν όσον αφορά τις επιβαρύνσεις και δεν θα είναι κάτι το οποίο θα δημιουργεί στρέβλωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να το δούμε αυτό. Οι προϋποθέσεις που θα δημιουργηθούν πρέπει να είναι βιώσιμες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Το πρόβλημα της χρήσης ε, των προϊόντων και τεχνολογιών που είναι πολιτικού χαρακτήρα για στρατιωτικό χαρακτήρα πρέπει να εξεταστεί και να δούμε ότι δεν εξαντλείται μέσα στο πλαίσιο των προϊόντων και ελέγχων τη χρήση. Είναι σημαντική αυτή η έλεγχη και πρέπει να γίνονται αποτελεσματικά και να μην ε, υπονομεύονται οι αναπτυσσόμενε χώρε για προϊόντα που έχουν ανάγκη να χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξή του. Πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια σε αυτό το πλαίσιο και να αυξηθεί ο δημοκρατικό έλεγχο. Αλλά και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι συνεκτική η Ευρωπαϊκή Ένωση με τι πολιτικέ που ακολουθεί σε σχέση με με τις προδιαγραφές αυτού του κανονισμού. Υπενθυμίζουμε προγράμματα ανάπτυξης υπό το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την ανάπτυξη με την συμμετοχή της αεροναυπηγικής βιομηχανίας του Ισραήλ και για την χρήση αυτών των προϊόντων στις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας που είχαν σαν αποτέλεσμα πάρα πολλά θύματα από πλευρά αμάχων. Και εδώ πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα προϊόντα διτής χρήσης που χρησιμοποιούνται με αυτόν τον τον τρόπο. Ευχαριστώ. Και τώρα για να κλείσουμε τη συζήτηση, πρώτα εξ ονόματο Επιτροπή η Επίτροπο η κυρία Μάλτστρομ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ισηγητά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος του κ. Ντεγκούχτ και σας και την Επιτροπή σας για το έργο σας. Συμμεριζόμαστε πολύ στις απόψεις σας στις εκθέσεις για τα δύο ζητήματα όπου ζητάτε εξάντε έγκριση. Είναι πάνω κάτω αυτό που θέλει και η Επιτροπή για να αποφεύγουμε τις πιθανότητες διπλών προδιαγραφών και τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε και έναν μηχανισμό εύκολων ε, εξαγωγών χωρίς να επιβάλλουμε μεγάλο άχθος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα όπου ελπίζω ότι θα βρεθούν ε, θα βρεθεί μια συμφωνία με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ εκ νέου για τη συζήτηση. μας ο κύριος Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τα τελευταία δύο λεπτά θα ήθελα να τα χρησιμοποιήσω για να απευθύνω μια έκκληση στο Συμβούλιο βλέπουμε κενά έδρανα εκεί που θα έπρεπε να είναι το Συμβούλιο. Και δεν είμαι βέβαιος αν θα πρέπει έτσι να διεξάγονται συζητήσεις ε, τη απουσία του Συμβουλίου. Σωστό θα ήταν να αναφερθεί στο Συμβούλιο ότι όταν επιθυμεί κάτι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προσέρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να παρακολουθεί τι συζητήσει στο σώμα αυτό και να δίνει απαντήσει. Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζω ότι είναι ένα μεγάλο οικονομικό τομέα αυτό. Πρόκειται για πολλά αγαθά, για θέσει απασχόληση για Ευρωπαίου και ιδιαίτερα για θέσει απασχόληση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι τεράστια σπουδαιότητα στο σύνολο της Ευρώπης πανευρωπαϊκά να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες και όχι να είναι δυνατόν μια χώρα να κάνει κάτι, μια άλλη να μην το κάνει και να έχει κάποιες διαφορετικές διατάξεις και πρακτικές. Δεν πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο. Γι' αυτό είναι σημαντικό εμείς να καταλήξουμε σε μια λύση του προβλήματος. Γοργά να επιλύσουμε το πρόβλημα και να δεχθεί επίσης το Συμβούλιο ότι δεν είναι δυνατόν όλα να γίνονται όπως τα φαντάζεται το Συμβούλιο. Είναι σημαντικό αυτό και αν αυτό γίνει αντιληπτό τότε μπορούμε γοργά να καταλήξουμε σε μια λύση που θα υιοθετηθεί προς το συμφέρον των ίδιων των πολιτών της Ευρώπης και της διασφάλισης της ασφάλειας και της δυνατότητας και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να τεθούν τα πράγματα σε τάξη. Αυτό ζητεί και η έκθεση. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λάκτριντ. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12. Το επόμενο σημείο σημερινής διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Σίμψον, Ευρωπαϊκές Στατιστικές στον τομέα του τουρισμού. Το λόγο έχει για τέσσερα λεπτά